με όλους τους ενδιαφερομένους και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι με την ανακοίνωσή μας αυτή. Σας ευχαριστώ. Κύριε και κύριοι συνάδελφοι, έχω λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος σχετικά με το θέμα της συζήτησης, επί των οποίων η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Το θέμα έληξε λοιπόν, η συζήτηση αυτή έληξε και ερχόμαστε στο επόμενο θέμα της ημερήσιάς μας διάταξης που προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις εισαγωγές κρέατος προέλευσης τρίτων χωρών. Θα ξεκινήσουμε με την Επίτροπο, την κυρία Βασιλείου. Έχετε το λόγο, κυρία Επίτροπο. Ε, να με συγχωρήσετε γιατί λόγω του θέματος αυτού που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολλές πτυχές θα μακρηγορήσω λίγο στην εισαγωγή μου προ όφελο των ε, εντύμων μελών του κοινοβουλίου. Ε, Αξιότιμα μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει πολλές ε, δέσμες κανόνων για τις εισαγωγές κρέατος προέλευσης τρίτων χωρών. Για σειρά ετών έχουμε μια πολύ αποτελεσματική πολιτική για τις εισαγωγές που λαμβάνει υπόψη τις επιστημονικές εξελίξεις και την κατάσταση των επιζωοτιών στις τρίτες χώρες. Ιδιαίτερα προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στον αυθόδη πυρετό στις χώρες από τις οποίες εισάγουμε διότι εμείς δεν έχουμε τέτοιου είδους κρούσματα και αν έχουμε θα υποστούμε πολύ σημαντικές οικονομικές συνέπειες. Είναι αυστηρές λοιπόν οι προϋποθέσεις και τα πρότυπα που ισχύουν σε επίπεδο των ε, διεθνών ε, οργάνων για την ε, μη εξάπλωση του αυτού του σπυρετού. Φυτικά και φυτογενομικά πρότυπα ε, μπορούν να είναι διαφορετικά και οι μέθοδοι διαφορετικές για την επιθεώρηση των προϊόντων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυξάνεται ο κίνδυνος για την ανθρώπινη αλλά και την υγεία των ζώων. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε ε, ένα ακριβές αντίγραφο των νομοθετικών μας προτύπων στις τρίτες χώρες. Όπως και οι τρίτες χώρες προς τις οποίες εμείς εξάγουμε δεν μπορούν να επιβάλλουν τους εθνικούς τους κανόνες σε εμάς. Εμείς μπορούμε μόνο να απαιτούμε ότι τα μέτρα τους έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα με τα δικά μας. Η ανιχνευσιμότητα. Ιδού ένα παράδειγμα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πολύ αυστηρούς κανόνες για την α, ταυτοποίηση και ανιχνευσιμότητα των βοηδών. Σε περίπτωση κρουσμάτων επιζωοτίας έχουμε ένα σύστημα ανιχνεύσης των ενδυνάμει ε, μολυσμένων ζώων για να σταματήσουμε την εξάπλωση της ασθένειας. Επίσης, οι κανόνες μας μας δίνουν τη δυνατότητα να ανοιχνεύουμε τροφές και ζωοτροφές καθόλη την διάρκεια της αλυσίδας, από τη φάρμα μέχρι το τραπέζι μας. Οι κανόνες ανιχνευσιμότητος ισχύουν λοιπόν και για τις τρίτες χώρες ακριβώς για να μην εκπροσωπεί κίνδυνο το εισαγόμενο κρέας. Βεβαίως αυτοί οι κανόνες έχουν πολύ πιο περιορισμένο βεληνικές από ότι στην Ένωση. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι τα μέτρα ενισχυσιμότητας των βοηθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίθηκαν μετά την κρίση της πογκόδους εγκεφαλοπαθίας που όπως θα ενθυμίστε ε, οδήγησε σε δραματική μείωση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των τιμών βεβαίως. Δράτω με τις ευκαιρίες για να εξηγήσω πιο λεπτομερώς τα μέτρα που έχουμε θεσπίσει για τις εισαγωγές βοήου κρέατος που διασφαλίζουν το υψίστο δυνατό επίπεδο προστασίας της ε, υγείας των καταναλωτών αλλά και των ζώων. ενώ συγχρόνω ε, ευθυγραμμιζόμαστε πλήρω με τα της συμφωνίας SPS. Είναι τόσο συνεκτικά που μόνο 12 χώρες εκτός Ευρώπης μπορούν να πληρώσουν όλα αυτά τα κριτήρια. Κατά συνέπεια, μόνο από αυτές τις 12 χώρες εισάγουμε κρέας. Πρώτον, οι εισαγωγέ βοηού κρέατο επιτρέπονται μόνο από τρίτε χώρε ή από ορισμένε περιοχέ τρίτων χωρών που έχουν ρητά εγκριθεί μετά από αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διαπιστώνει ότι τα πάντα έχουν καλώς. Δεύτερο, η περιοχή προέλευσης πρέπει να χαρακτηρίζεται από την ΟΑΗ e και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ελεύθερη επιζωτιών και ιδίως αυτό το Δι, ε, τρία. Το εισαγόμενο κρέας πρέπει να συνοδεύεται από ένα συγκεκριμένο σχέδιο και πρόγραμμα ε, για κατάλοιπα από κτηνιατρικά προϊόντα, από ορμόνες που απαγορεύονται ή μπορούν να ε, χρησιμοποιούνται μόνο περιορισμένα. Τέταρτο, όλες οι εισαγωγές νοπού κρέατος προέρχονται από διαπιστευμένο συμβεβλημένο σφαγείο. 5. Υπάρχουν ιδιαίτερα πρότυπα για την παραγωγή και αποθήκευση του κρέατος. Έχουμε άλλο ένα στρώμα μέτρων που αφορούν τι αγωγές από την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Χιλή, τη Νέα Ζηλανδία και τι Ηνωμένες Πολιτείες. Για τι 7 υπόλοιπες εξοδοτημένε χώρες μόνο αποστεωμένο κρέα μπορεί να εξαχθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι διασφαλίζουμε την αδράνεια του ιού ακόμα και αν υπάρχει μετά την εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων. Πρόκειται λοιπόν για ένα περαιτέρω δίκτυο ασφαλείας. Οι παρτίδε του κρέατο που πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί από επίσημο κτηνίατρο που εγγυάται ότι όλες οι προϋποθέσεις που ανέφερα προηγουμένως πληρούνται. Όταν φτάνει η παρτίδα στην Ένωση γίνονται έλεγχοι από τι επίσημε κτηνιατρικές αρχέ των κρατών μελών στις στα σημεία ελέγχου στα σύνορα. Όλο το εισαγόμενο κρέας πρέπει να υποστεί υποχρεωτικούς ελέγχους στα σύνορα. Στο συνοριακό φυλάκιο, στα τελωνία, γίνεται ταυτοποίηση της προέλευσης, φυσική έλεγχη, αλλά και έλεγχη των συνοδευτικών εγγράφων. Επιπροσθέτως, γίνεται και φυσικός κτηνιατρικός έλεγχος. Κατελάχιστον 20% όλων των παρτίδων εισαγωμένου κρέατος. Και υπάρχει κι άλλο ένα επίπεδο προστασίας, πρόσθετο, λόγω της απαγόρευσης ορισμένων πρακτικών για την εισαγωγή κρέατος στην Ένωση. Ορισμένα είδη ευάλωτα στην Ένωση δεν μπορούν έτσι να εκτεθούν στον ιό της επιζωοτίας αυτής ακόμα και αν αυτός επιζήσει παρά τα μέτρα που περιέγραψα. Μέτρα που είναι πλήρως συναρμονισμένα. Το 2006 η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιστημικής Ασφάλειας ανεγνώρισε ότι τα μέτρα αυτά είναι πολύ αποτελεσματικά για την μείωση της, ε, των ε, κινδύνων εισαγωγής της ασθένειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι και κατά λέξη παραθέτω απέδειξε ότι έχει ένα ε, πολύ αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου. Τα μέτρα αυτά λοιπόν είναι αποτελεσματικά για το εμπόριο προϊόντων κρέατος και νοπού κρέατος. Φτάνω έτσι στο επόμενο σημείο. Από την εναρμόνιση των ε, κανόνων στα κτηνετρικά τη δεκαετία του 70 ποτέ δεν υπήρξε ε, επιδημία της συγκεκριμένης επιζωτίας μέσω των νομίμων εισαγωγών. Να μην ξεχνάμε ότι ο αυθόδης πυρετός το 2001 στην Ένωση προκλήθηκε από την παράνομη εισαγωγή κρέατος, μάλλον από την Ασία, και ε, την παράνομη χρήση ζωοτροφών για τους χείρους. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε που έγκυται ο κίνδυνος και να στοχοθετήσουμε σωστά τα νομοθετικά μας μέτρα και τα μέτρα ελέγχου. Είδατε τις αφήσει στα αεροδρόμια της Ένωσης και σε άλλα σημεία εισόδου που εξηγούν στους ε, ταξιδιώτες τους κανόνες που αφορούν την εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης. Γνωρίζω ότι ορισμένοι εξημών έχετε εκφράσει ανησυχίες για το βόλιο κρέας που εισάγουμε από τη Βραζιλία. Σας παραπέμπω στους κανόνες που εγκρίναμε πέρσι το Γενάρη. Κανόνες που περιλαμβάνουν πέρα από όλα αυτά που ανέφερα ήδη την υποχρέωση να έχουν εγκριθεί από τις βραζιλιανές αρχές τα ζώα αυτά των οποίων το κρέας όταν έχει προέλευση την έχει ε, προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σε μια βάση δεδομένων. Τα ζώα αυτά είναι λιγότερο από το 1,5% της συνολικής βραζιλιανής ε, του συνολικού πληθυσμού που είναι 2,9 εκατομμύρια κεφάλια. Κατά συνέπεια οι βραζιλιανές αρχές κάνουν νέε αξιολογήσει των εκμεταλλεύσεων που θέλουν να παράγουν κρέα για εισαγωγή στην Ένωση. Από πάνω από 10.000 εκμεταλλεύσεις επιλέξιμες το Νοέμβριο του 2007 ήταν μόνο 1.708. Κατά συνέπεια, οι εισαγωγές βραζιλιανού βοήου κρέατος έχουν μειωθεί κατά πολύ. Αρχές του 2009 εντοπίστηκαν κάποια ελλείμματα κατά μια επιθεώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι Βραζιλιανές χερσές επέδειξαν πλήρη συνεργασία για να ε, ρυθμίσουν το πρόβλημα. Πάντως, τα συνολικά αποτελέσματα δεν δικαιολογούν περαιτέρω περιορισμούς των εισαγωγών του βραζιλιανού βοηού κρέατος στην Ένωση. Ισότι αφορά το πώς έχουν τα πράγματα τώρα. Η επιβολή νέων περιορισμών για την εισαγωγή βοήου κράτου από τη Βραζιλία θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως προστατευτισμός από ορισμένους και θα μπορούσε να οδηγήσει σε προσφυγή σε πάνελ του ΠΟΕ. Πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από καιρού εις καιρών έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα δικά μας προβλήματα. Και θέλουμε να αντιδρούμε κατά αναλογικό τρόπο. Θα πρέπει να δίδουμε το παράδειγμα και να ακολουθούμε τους κανόνες που διέπουν το διεθνές εμπόριο. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να ε, στοχοθετεί τις προσπάθειές της στις παράνομες εισαγωγές που αυτές είναι η πηγή κινδύνου. Θα διατηρήσουμε επίσης την υφιστάμενη αναλογική μας αντιμετώπιση των εισαγωγών από τρίτες χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Βραζιλίας. Αυτό θα διαβεβαιώσει, θα διασφαλίσει ότι έχουμε υψηλά επίπεδα προστασίας ε, ανθρώπινης υγείας και υγείας των ζώων αλλά και ότι θα έχουμε αξιοπιστία σε διεθνές επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ε, και το λόγο τώρα θα, θα πάρουν οι βουλευτές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Εράνς για δύο λεπτά εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει στους κοινοτικούς παραγωγούς πολύ αυστηρά πρότυπα, πολύ αυστηρότερα από αυτά που υπάρχουν σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί υποχρεούνται να πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις γιατί αλλιώς δεν λαμβάνουν ενίσχυση για τους περισσότερους δεν αξίζει τον κόπο οικονομικά. Είναι ηλικιώδης ο ρυθμός εγκατάλειψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Αν δεν λάβουμε μέτρα, οδεύουμε προς την καταστροφή. Τέλος πάντων, το έλλειμμα της Ένωσης καλύπτεται το συνολογικό από, από εισαγωγές τρίτων χωρών, με επικεφαλής την Βραζιλία. Είναι έλλειψη ειλικρίνειας να αφήσουμε να περάσουν στην Ένωση παρτίδες κρέατος που δεν πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα που έχουμε θεσπίσει. Πρότυπα που είναι χαμηλότερα από αυτά που ισχύουν για τους δικούς μας παραγωγούς. Διότι από ό,τι φαίνεται να επιβάλλουμε τους ακριβώς ίδιους κανόνες θα ήταν κατά των όσων ισχύουν στον ΠΟΕ. Αλλά αφού ο ΠΟΕ δεν μας το επιτρέπει αυτό, να έχουμε τα ίδια επίπεδα δηλαδή προτύπων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τουλάχιστον θα έπρεπε να διασφαλίσει ότι όλο το κρέας που περνά τα ευρωπαϊκά σύνορα προέρχεται από εκμεταλλεύσεις που έχουν υποστεί αν μη τι άλλο τον κατάλληλο έλεγχο. Η ζήτηση είναι αρκετή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα εθελοτυφλούμε και ότι θα παραβλέπουμε τις ατασταλίες που μπορεί να ανοιχνεύσουν οι κοινοτικές υπηρεσίες στις επιθεωρήσεις που κάνουν ερώτημα. Γιατί πάση θυσία προσπαθεί η Κομισιόν να ελαχιστοποιήσει τα προβλήματα αυτά. Ενώ είναι γνωστό ότι πολλά πιστοποιητικά από τη Βραζιλία δεν γίνονται σωστά. Έχουν εντοπιστεί πολύ μεγάλα προβλήματα στο σύστημα ανιχνευσιμότητας αυτής της χώρας και έχουν ανιχνευτεί προβλήματα με πολλές παρτίδες που δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικά. Πώς μπορείτε να διασφαλίσετε ότι οι 1.500 βραζιλιανές εκμεταλλεύσεις πληρούν τις προϋποθέσεις για τις οποίες έχει υπογραφεί η συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ, αλλά μην ξεπερνάτε το χρόνο κύριοι συνάδελφοι. Ο κύριος Κέλλη για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Uh, thank you, President. When it... Ευχαριστώ. Όσον αφορά το ζήτημα των εισαγών κρέατος, εμείς πρέπει να θέσουμε την πολιτική, να υπάρχει ένα δίκαιο σύστημα ε, κανόνων. Οι αρχές πρέπει να βασίζονται στην ασφάλεια των καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος, ε, την εμπιστοσύνη και ισότιμη μεταχείριση των παραγωγών κρέατος. Αυτή τη στιγμή το σύστημα ουσιαστικά είναι άνισο και για τους γεωργούς ε, και για τους καταναλωτές ε, είναι πάρα πολύ δαπανηρές οι πρακτικές ε, και τελικά εισάγουμε κρέας ε, από άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως από την Βραζιλία. Αυτή η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη. Οι πρακτικές στη Βραζιλία ε, σε μερικές ε, περιπτώσεις ε, δεν πληρούν προδιαγραφές που να είναι αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα εξαφανιστεί το ποιοτικό κρέας αν επιτρέπουμε να αποδυναμώνεται το εισόδημα των παραγωγών με τέτοιο τρόπο. Επίσης, έτσι όπως είναι η αλυσίδα η διατροφική, από τη στιγμή που υπάρχει το κρέας και πηγαίνει από τη μία χώρα στην άλλη, δεν είναι όλα αντικείμενο ανιχνευσιμότητας ειδικότερα για το βοδινό κρέας. Ε, και το αποτέλεσμα βέβαια είναι αρνητικό για τους καταναλωτές. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι τα νέα μέτρα ε, είναι τα κατάλληλα και υπάρχουν πάρα πολλά ε, παραδείγματα σε πολλές περιπτώσεις θεωρούνται εγκεκριμένε εκμεταλλεύσεις που δεν είναι εγκεκριμένε όμως. Νομίζω ότι έχει φτάσει η στιγμή να αντιδράσουμε. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η πρακτική. Είναι άδικη για τους καταναλωτές, είναι άδικη για τους παραγωγούς, είναι άδικη για τους παραγωγούς στην Ευρώπη που έπρεπε να ακολουθήσουν πρακτικέ οι οποίες ε, δεν ε, είναι αποδεκτές από τις ε, Απραγού Βραζιλία. Λίον, έχει το λόγο για δυόμιση λεπτά παρακαλώ, την ομάδα των φιλελευθέρων. Ε, thank you, ε, President, and thank you, Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστούμε και την Επιτροπή για τη δήλωσή τη Η γκάμα των μέτρων προστασίας που ανελήφθησαν πραγματικά είναι ε, και χρήσιμη. Να πω μερικά πράγματα τώρα σχετικά με το κρέας που έρχεται από τη Βραζιλία. Η μέθοδοι ανιχνευσιμότητας και η δυνατότητα τα μέτρα σχετικά με την ανιχνευσιμότητα πρέπει να είναι κύρια στο σύστημα που έχουμε για την εισαγωγή προϊόντων κρέατος από τη χώρα αυτή για να ελεγχιστοποιήσουμε τους κινδύνους για τους πολίτες κοινότητας. Πα, παρόλα αυτά υπάρχει πρόβλημα. Η έκθεση της ε, Κομισιόν το Φεβρουάριο μας είπε ότι 50% των ε, κτηνοτρόφων ε, που ελέγχθησαν και για να πάρουν έγκριση για εξεγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν προβλήματα για πάρα πολλά προϊόντα δεν ξέραμε από που προέρχονταν δεν υπήρχαν τα σχετικά έγγραφα ένας από τους κυβερνητικούς επιθεωρητές δεν έκανε καλά τη δουλειά του και μάλιστα ήταν και ιδιοκτήτης του ζωικού κεφαλαίου των, ζώων και της φάρμας από την οποία είναι σε οι και παρόλα αυτά το αποτέλεσμα στο έγγραφο ήταν ότι όλοι οι έλεγχοι ήταν ικανοποιητικοί. Αυτό δεν αρκεί. Πιστεύω ότι πρέπει να επαγρυπνούμε όλοι μας όντως η εμφάνιση μιας κάποιας νόσου όπως η οφθόδης πυρετός θα έχει τεράστιες συνέπειες και οικονομικές και άλλες στην ε, Αγγλία κόστισε η υπόθεση αυτή τέσσερα δις στερλίνες και αναγκαστήκαμε να θανατώσουμε πάρα πολλά ζώα δεν ζητώ να επιβάλλουμε ε, τους δικούς μας κανόνες στη Βραζιλία. Ζητώ όμως απόψε να επαγρυπνούμε, να κάνουμε καλούς ελέγχους και η επόμενη έκθεση από τους ελέγχους αυτούς να είναι πραγματική ούτως ώστε να μπορούμε να είμαστε ήρεμοι για τις εισαγωγές από τη Βραζιλία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σμίθ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πολύ ε, πλήρη δήλωση την οποία μας κάνετε και η οποία πραγματικά ήταν εξαιρετική. Ελπίζω η παρουσία των μελών εδώ απόψε τόσο αργά να σας πείθει για το γεγονός ότι ενδιαφερόμαστε για το θέμα καταλαβαίνουμε την απειλή και τους κινδύνους που προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε εσείς σχετικά με τον αυθόδη πυρετό το πρόβλημά όμως δεν είναι η οι επιζωτίες δεν είναι καν οι εισαγωγές από τη Βραζιλία. Οι ψηφοφόροι μας ζητούν γενικώ αυτοί οι οποίοι εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόν, να έχουν τα ίδια στάνταρτ, τα ίδια πρότυπα που έχουμε και εμείς. Και αυτό βεβαίως ε, και αυτό ακριβώς περιμένουν οι οι ε, πολίτε μα θέλουν ακριβώ τα ίδια πρότυπα να εφαρμόζονται. Καταλαβαίνω αυτό που είπατε εσεί. αλλά θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, οι πολίτε μας και οι αγρότε μας και εμεί ζητούμε ακριβώ τα ίδια στάνταρ χνηλασιμότητας όπως ανιχνευσιμότητας όπως ισχύουν και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουμε να προκαλέσουμε τα πράγματα. Θα θέλαμε γι' αυτό να μας πείτε πότε θα υποβάλλετε την επόμενη έκθεσή σας και πότε τέλος πάντων θα απαγορεύσετε τις εξαγωγέ από τις χώρες που δεν τηρούν τα ευρωπαϊκά στάνταρτς. Νίκολσον, κυρία Πρόεδρε, Πρώτα πρώτα να πω ότι η συζήτηση εδώ δεν η σχετίζεται γενικώ με τις εξαγωγές τρίτων χωρών όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε ειδικά για το κρέας που έρχεται από τη Βραζιλία και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έχουμε ψήφισμα, γιατί οι πολιτικές ομάδες αυτού του κοινοβουλίου δεν μπόρεσαν να φτιάξουν ένα ψήφισμα κοινό για να ε, αντιμετωπίσουμε τη Βραζιλία. Θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι οι Βραζιλιάνοι δεν με πίεσαν, δεν ήρθε το λόμπι το βραζιλιάνικο σε μένα ή γιατί πιστεύουν ότι δεν άξιζε να το κάνουν ή γιατί θεώρησαν θα είμαι πολύ σκληρός και λέω απόψε κυρία Επίτροπε εσείς και η Κομισιόν δεν μπορείτε να δέστε τα χέρια των Ευρωπαίων αγροτών και να τους αναγκάζετε να ε, εφαρμόζουν standards πανδύσκολα όταν δεν κάνετε το ίδιο και για άλλες χώρες. Δεν ξέρω κύριε Επίτροπε πόσα χρόνια θα μείνετε, δεν ξέρω ποιος θα σας αντικαταστήσει αλλά αυτό που λέω θα το επαναλάβω και στους διαδόχους σας το στάνταρ του κρέατος που έρχεται στην Ευρώπη πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που παράγουμε. Δεν πρόκειται να υποκύψουμε, να συνεχίσουμε να υποκύπτουμε ε, σε χαμηλή ποιότητα κρέατα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νικόλσον. Ο κύριος Μπάφτον για δύο μισή λεπτά παρακαλώ. Um, Ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να αναφέρω κάποιες σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα του κρέατος από τη Βραζιλία. Ε, το κρέας αυτό μπορεί να είναι μολυσμένο από τον αυτό διπηρετώ όπως ακούσαμε και το ότι δεν υπάρχουν κανόνες στη Βραζιλία σημαίνει ότι οι κτηνοτρόφοι εκεί έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους Ευρωπαίους κτηνοτρόφους και περαιτέρω πρόβλημα υπάρχει και λόγω της κλιματικής αλλαγής κλιματικές αλλαγές η Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνει τόσα πράγματα για την κλιματική αλλαγή γιατί ε, αγνοείται ότι η Βραζιλία καταστρέφει το, τα τροπικά δάση τα παρθένα δάση το 80% των παρθένων δασών όλ, καθημερινά όλο και πιο πολλά αγροκτήματα και εκτινοτροφικές εκμεταλλεύσεις εγκρίνονται για να εξάγουν κρέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες σχετικά και για τις εκμεταλλεύσεις και για τα σφαγεία και ε, για την ε, τους ελέγχους που γίνονται πριν δοθούν οι εγκρίσεις και οι εξουσιοδοτήσεις. Εμείς εδώ στην Ευρώπη πρέπει να προστατεύσουμε εκτός από τους κτηνοτρόφους και τους καταναλωτές μας. Η κτηνοτροφία στην, Ευρώπη στην Ευρώπη αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό από τους παραγωγούς εκτός Ευρώπης πολλές αλυσίδες καταστημάτων όπως η Walmart και το Carrefour απαγόρευσε δεν πουλάει πια ε, κρέας από τη Βραζιλία και ε, η κτηνοτροφία στη Βραζιλία όπως σας είπα καταστρέφει το 80% των τροπικών δασών είναι κάτι που δεν μπορούμε να το δεχτούμε και δεν πρέπει να το δεχτούμε ως Ευρώπη. Πολύ κύριε Μπάφτον. Ε, θέλετε, μπορεί να σας υποβάλει μια ερώτηση, Mr. Μπάφτον. Μπορείτε να σας υποβάλει μια ερώτηση ο κύριος Σμιτ. Θέλετε ο κύριος Σμιτ να σας υποβάλει μια ερώτηση, θέλει να κάνει χρήση του δικαιώματος blue card. Yes. Mr. Smith, you have the floor. Uh, ευχαριστώ Καταλαβαίνω αυτά που είπε ο κύριος Πάφτον, αλλά θα ήθελα να τον ρωτήσω κάτι. Είπε ότι το κρέας ε, που δεν ελέγχεται σωστά ε, εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή ακούσαμε και μία παρουσίαση από την Επίτροπη πριν από λίγο, από ό,τι κατάλαβα δεν ισχύει αυτό και μήπως υπερβάλλεται λιγάκι και το θέμα ολόκληρο αποδυναμώνεται, όλη η συζήτηση αποδυναμώνεται γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ τεχνικό κείμενο, νομοθετικό και δεν νομίζω ότι βοηθάτε την κατάσταση. Αντιθέτω παρακολύεται. Ναι, βεβαίω να απαντήσω. Αν δούμε τι συμβαίνει με, τις, με το εισαγόμενο κρέα από τη Βραζιλία, για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Ναι, δεν ε, ισχύουν οι κανόνε για το συγκεκριμένο κρέα. Αυτό υπάρχει. Αυτό που είπατε είναι μεν πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να σα πω ότι υπάρχει τέτοιου είδου κρέα που εισάγεται από τρίτε χώρε και αν δεν είμαστε... Ε, αφού δεν είμαστε προσεκτικοί, προέκυψε η κατάσταση που έχουμε. Γιατί για ποιο λόγο μιλάμε τότε για μη ελεγχόμενο κρέας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν υπάρχει το πρόβλημα που ανέφερα. Προφανώς υπάρχει το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Bafton. Ε, ε, και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ντότζ για ένα λεπτό. Ε, Πρόεδρε, Επίτροπε, ευχαριστώ. Όπως πολλά από τα εδώ περιστάμενα μέλη, τελώ σε σύγχυση με την αποδοχή σας ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τις εισαγωγές κρέατος από τις χώρες του τρίτου κόσμου, του, από τρίτες χώρες, Λέτε ήδη από την αρχή της παρέμβασής σας ότι όπως εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε σε αυτούς και αυτοί δεν μπορούν να επιβάλλουν σε εμά. Ή μάλλον εφόσον αυτοί δεν μπορεί να επιβάλλουν σε εμά και εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε σε αυτούς. Δεν είναι σωστό. Ε, μπορούμε να επιβάλλουμε. Μπορούμε να επιβάλλουμε κανόνες μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι τα πράγματα έχουν καλώς. Μέχρι η κτηνιατρική δεν μπορουν να πιστοποιούν πράγματι ότι οι τρίτες χώρες συμφωνούνται ε, συμμορφούνται συγγνώμη, με τους ε, κανονισμούς που ισχύουν στην Ένωση. Σε αντίθετη περίπτωση να μην εισάγουμε. Πολλέ χώρες υποφέρουν ε, από την κατάσταση αυτή και νομίζω ότι ακούτε το θυμό που έχουν πολλοί συνάδελφοι για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Αντότ. Συνεχίζουμε τον κατάλογο με τους άλλους εγγεγραμμένους ομιλητές. Η κυρία Μαγκίνες για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως ε, συνσυντάκτρια αυτής της ερώτησης, συμφωνώ και δακτυλοδεικνύω τους σοσιαλιστές που χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για πολιτικούς ή πολιτικάντικους λόγους. Ευχαριστώ Επίτροπε για την ε, λεπτομερή σας ε, παρουσίαση αλλά νομίζω ότι δεν είπατε το πιο βασικό ότι λάβατε δράση μόνο λόγω δράσης που ανέλαβαν οι Ιρλανδοί γεωργοί μετά από δική μας εισήγηση. Πολιτική πίεση είναι αυτή που σας ανάγκασε να αναλάβετε δράση. Εγώ σημείωσα τα όσα είπατε και θα ξαναδιαβάσω όλη σας την ομιλία αλλά θέλω να το αποδεχτείτε αυτό ότι σας ανάγκασαν οι πιέσεις να αναλάβετε δράσεις. Το 2007 10.000 επιλέξιμες εκμεταλλεύσεις. 1.700 σήμερα. Τι μου λέει εμένα αυτό? Ότι οι υπόλοιπες 8.300 δεν θα έπρεπε να έχουν καν εισάγει μία φορά, εξάγει μάλλον, μία φορά κρέας προς την Ένωση. Δύο τινά δεν εμπιστεύομαι την υφιστάμενη Επιτροπή να αντιμετωπίσει υπεύθυνα και αποτελεσματικά το πρόβλημα. Την επόμενη Επιτροπή, τα μέλη και τον πρόεδρο της επόμενης Επιτροπής προειδοποιώ ότι θα το, θα το πάμε μέχρι τέλους τον αγώνα μας. Να υπάρχουν υψηλά πρότυπα παντού. Αν μειωθούν τα πρότυπα αυτά λόγω ατασταλιών από εισαγωγές από τρίτες χώρες, θα υποστείτε τις συνέπειες του θυμού που υπάρχει στην κοινότητα των γεωργών και κτηνοτρόφων στην Ένωση. Να είστε σίγουροι, Επίτροπε. Μπορεί να είναι αργά, αλλά είμαστε ξύπνοι. Ευχαριστώ κύριε Μακίνες. Ο κύριος Ταραντέλα για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, ποια είναι η διαφορά μεταξύ της του ευρωπαϊκού κρέατος και του κρέατος από τη Βραζιλία. Δεν είναι τόσο η γεύση, είναι οι διαφορετικοί κανόνες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχουν υποχρεωτικά στις τρίτες χώρες από τις οποίες εισάγουμε το κρέας. Για παράδειγμα, για το κρέας της Βραζιλίας, ε, όπου στις οποίες αναφερθήκατε κι εσείς ε, για τους ελέγχους τους κτηνιατρικούς σε μια έκθεση που μας υποβάλλατε το 2007. Επίσης φάνηκε ότι η βακτηριολογική ποιότητα του αργεντίνικου κρέατος ήταν χαμηλότερη από, την τοπική, από το τοπικό κρέας ε, και αυτό δεν είναι εκπληκτικό αν ε, δούμε ότι χρειαζόμαστε δύο μήνες για να έρθει το κρέας από την Αργεντινή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως η κατανάλωση είναι πολύ πιο σύντομη. Για παράδειγμα στο Βέλγιο ε, γίνεται η κατανάλωση εντός του μηνός από τη σφαγή. Γιατί, γιατί αυτό ακριβώς ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λέμε ότι πρέπει να το υποβάλουμε σε τρίτες χώρες, αλλά πρέπει και οι τρίτες χώρες που εξάγουν ε, κρέα σε εμά να δέχονται τους κανόνες μας διαφορετικά. Για ποιο λόγο τότε λέμε ότι δεν υπήρξε ε, προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με τη Χιλή και με τη Βραζιλία έχουμε δείξει πώς πρέπει να κινηθούμε, ε, γιατί εμείς απαγορεύσαμε τουλάχιστον τις εισαγωγές του κρέατος και νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος να εξασφαλίσουμε την ποιότητα. Η κυρία Χόρκιν έχει το λόγο. Thank you, Madam Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, Είπατε ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τις ίδιες, τους ίδιους κανόνες, αλλά πρέπει να έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα. Μιλήσατε για την ανιχνευσιμότητα από τη φάρμα στο πιάτο μας, αλλά μας είπατε επίσης ότι σε τρίτες χώρες ε, η ανιχνευσιμότητα είναι πολύ πιο περιορισμένη. Αν λοιπόν ισχύει αυτό, και αυτές ήταν οι, δική σας λέξη, οι δικές σας λέξεις, πώς μπορούν να έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα. Το θέμα είναι το εξή. Η πρόσφατη έκθεση του ΦΑΟ για την εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία. Το πρόβλημά μου είναι το εξή. Και η Κομισιόν και ο ε, πάρα πολλές φορές ε, υποτίμησαν τα πορίσματα των μελετών τους. Ναι, όντως υπήρξαν κάποια επιπλέον, κάποιες επιπλέον ε, απαιτήσει, αλλά όπως είπε και η συνάδελφος υπήρχε πάρα πολύ μεγάλες, μεγάλη πίεση από την Επιτροπή Γεωργίας εγώ ε, αν έδινα στους φοιτητές μου 12 ε, ασκήσεις να κάνουν και μόνο 6 λύνανε, ε, τι να σας πω, ε, δεν θα παίρνανε καλή βαθμολογία, δεν θα το θεωρούσε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, ειδικότερα αν πάρα πολλά χρόνια προσπαθούσα να τους βοηθήσω να βελτιώσουν την επίδοσή τους. Καλό είναι το ελεύθερο εμπόριο, αλλά και οι Ευρωπαίοι καταναλωτές χρειάζονται ασφάλεια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο πρέπει να εξασφαλίσουν και τα δύο. Εγώ δεν θα τους έδινα και καλό βαθμό για τη δουλειά του. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άσγουρθ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, χάρηκα που είστε αποφασισμένοι να διατηρήσετε ψηλά στάνταρ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ήθελα να πω το εξή. Μιλήστε για τις αφήσει στα αεροδρόμια. Οφείλω να σας πω ότι δεν είδα καμία προειδοποίηση, καμία, κανένα έλεγχο να γίνεται στα αεροδρόμια, στα εισαγόμενα προϊόντα. Οπότε ξανακοιτάξτε το γιατί νομίζω ότι δεν έχετε δίκιο. Δεύτερο, δεν είμαι πεπισμένος για αυτά που είπατε για το κρέας από τη Βραζιλία. Πήγα στην ε, Βραζιλία και είδα τα πράγματα επί τόπου και υποστηρίζω πολλά από αυτά που ελέγχθησαν. Οι κτηνοτρόφοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίνονται σε πολύ ψηλά στάνταρτ, κυρία Επίτροπε, και αυτό κοστίζει ένα κόστος, μιλάμε ένα κόστος που δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε στους ε, καταναλωτές μας. Οπότε δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ούτε από τους αμπεκτηνοτρόφους ούτε από τους καταναλωτές ένα προϊόν το οποίο είναι ε, χαμηλότερης ποιότητας ή δεν έχει περάσει από κάποιους ελέγχους δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο και αυτό δεν είναι προστατευτισμός είναι η εφαρμογή κοινή αγροτικής πολιτικής που θα έπρεπε να προβλέπει παροχή καλού, το, καλών διατροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και ασφαλών Δες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε Κυρία Επίτροπε Ευχαριστώ την κυρία Χέρανς που έφερε εδώ σήμερα στο Κοινοβούλιο το θέμα αυτό γιατί αυτό που συζητούμε είναι βασικότατο θέμα στον τομέα των τροφίμων. Εγώ δεν ενδιαφέρομαι ε, να ε, επικρίνω τη Βραζιλία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι κατά πόσο ο Ευρωπαίος καταναλωτής χρειάζεται απαραίτητο σε αυτές τις εισαγωγές. Αν ε, η απάντηση είναι ναι, τότε ρωτώ. Α, δεν πρέπει να προστατευθεί ο, ο καταναλωτής και αυτό σημαίνει περισσότερο κόστος που αναλαμβάνουν οι δικοί μας παραγωγοί αλλά όχι αυτοί σε τρίτες χώρες δεν είναι δυνατόν να ε, τιμωρείται ο Ευρωπαίος κτηνοτρόφος σε κάποιο έλεγχο γιατί ο δειγματοληπτικός έλεγχος έδειξε να έχει γίνει ένα λάθος όταν κατακλυζόμαστε από εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει ασφάλεια των εισαγωγών και προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών έχω την εντύπωση ότι οι υπεύθυνοι για τις ε, εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιούν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ε, εγώ δεν θέλω να ε, ε, περιχαρακωθούμε μέσα σε ένα οχυρό Ευρώπη και να απομονωθούμε. Όχι, θέλω όμως οι πολίτες της Ευρώπης να είναι ασφαλείς και ε, να προστατεύονται και σας λέω απλώς κυρία Επίτροπε ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να θέτει το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων και για την, ε, τον διάδοχο και ενώπιον του διαδόχου σας ενώπιον της νέας ε, Κομισιόν. Ο κύριος Κορτές Λάστρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Sí, Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι, πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να εξασκεί, να ασκεί έλεγχο για τις εισαγωγές από τις τρίτες χώρες. Είναι υποφελές για όλους, και τους ε, Ευρωπαίους παραγωγούς και τους καταναλωτές που ε, ζητούν ποιοτικά αγροτικά προϊόντα που να πληρούν τις προϋποθέσεις για την ευημερία των ζώων και την αλλά και στι τρίτε χώρε που θέλουν να εξάγουν τα προϊόντα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλο, θα ήθελα να επιθυμήσω ότι το πρόβλημα αυτό δεν περιορίζεται μόνο στον τομέα μια χώρα. Το θέμα τη ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γενικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκίρλιν έχει το λόγο για ένα λεπτό. Thank you, Madam President. My region of the southwest of England is blessed. Στην περιοχή μου, στην ε, νότιο Δυτική Αγγλία έχουμε πάρα πολύ ε, καλό κλίμα και ε, πολύ καλή κτηνοτροφία και παράγουμε πάρα πολύ καλό κρέας. Αυτό είναι σημαντικό να το σημειώσετε με δεδομένο ότι αυξάνεται ο πληθυσμό της γης και η κατανάλωση κρέατος θα έπρεπε η κτηνοτρόφοι της περιοχής αυτής να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι αλλά υπάρχουν και οι φυτοφάγοι οι, αυτοί που δεν τρώνε κρέας όπως μας είπα προηγούμενα συνάδελφος και φαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο υποστηρίζει αυτή την προσέγγιση από την άλλη μεριά εισάγουμε κρέας από περιοχές που καταστρέφουν τα δάση ε, τους λόγου για να παράγουν το κρέας αυτά είναι παράδοξα πράγματα δεν είναι ικανοποιημένοι ούτε κτηνοτρόφοι ούτε οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ζητώ κυρία Επίτροπε να τα προσέξετε ιδιαίτερα σε αυτά. Ο Λαβία έχει το λόγο τώρα για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, πιστεύω ότι το θέμα το οποίο συζητούμε απόψε είναι ένα μικρό κομμάτι ενός πολύ μεγαλύτερου προβλήματος. Η ισότιμη συμπεριφορά μεταξύ αυτών που επιβάλλουμε στους γεωργού μας και αυτό που δεχόμαστε από τρίτους δεν αφορά μόνο τις αγωγές κρέατος αλλά και πολλά άλλα α, προϊόντα. Εις ό,τι αφορά το κρέας, είμαστε καθαρός εισαγωγέας μόνο το 60% των αναγκών μας παράγουμε. Είμαστε αναγκασμένοι να εισαγάγουμε λοιπόν. Αλλά θέλουμε να προστατεύσουμε και τους καταναλωτές. Θέλουμε η υγεία να την χάνει προστασίας παντού στην Ένωση αυτό που είπατε σήμερα, ότι δεν είναι δυνατό να επιβάλλουμε ανάλογες συνθήκες εισαγωγής στις τρίτες χώρες, θέλουμε να μην το ξανακούσουμε ποτέ. Ποτέ. Δεν είναι αυτός ο δρόμος που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Η ανιχνευσιμότητα του προϊόντος η ισοτιμία των προτύπων που ισχύουν εδώ και αλλού είναι πολύ σημαντικές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λαβία. Η κυρία Ντελόγκε για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι η τελευταία ομιλήτρια και θα προσπαθήσω να συνοψίσω. Νομίζω ότι μπορώ να το κάνω. όλοι μας Όταν θέλουμε να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση πρέπει να σεβόμαστε και τους ίδιους κανόνες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν λοιπόν οι κανόνες δεν είναι ίδιοι, οι κανόνες δεν είναι ίδιοι για όλους, τότε οι παραγωγοί μας ε, θα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν ε, στους διεθνείς ε, κανόνες. Και αυτό ισχύει και για το εισαγόμενο κρέας ε, από τη Βραζιλία και για πολλά άλλα πράγματα. Δεν χρειάζεται να σα τα απαριθμίσω. Όταν σας ακούω, έχω λίγο την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε Μερικέ φορές να μην ισχύουν όλοι οι κανόνες, ε, να μην ισχύουν με τον ίδιο τρόπο οι κανόνες για όλους. Βεβαίω έχει σημειωθεί πρόοδο ω προ τον εμβολιασμό και ω πολλά, ε, πολλά τέτοια θέματα ε, η δική, μας, η δική μου χώρα έπρεπε να σφαγιάσει πάρα πολλά ζώα επειδή υπήρχε κρίση η επιζωτία του αυθόδου σπυρετού. Αλλά πρέπει και οι τρίτες ε, χώρες να μπορούν να σέβονται τις ίδιους κανόνες. Τώρα είμαστε στη διαδικασία Catch the Eye και ήδη έχουν ζητήσει το λόγο αρκετοί συνάδελφοι. Ο, ο κύριος Γιάχρε έχει το λόγο πρώτος. Για ένα λεπτό παρακαλώ, μην ξεπεράσετε το χρόνο. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ειδική στα κτηνοτροφικά και αγροτικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουν πει επανειλημμένα ότι ό,τι ισχύει στο εσωτερικό πρέπει να ισχύει και για τις εισαγωγές με μεγάλη ε, προσοχή παρακολούθησε την κυρία Επίτροπο η οποία επί 10 λεπτά προσπαθούσε να μας πει γιατί κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύει Νομίζω ότι εκείνο που επιθυμούμε εμείς, τουλάχιστον η δική μου πολιτική ομάδα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Εκείνο που επιθυμούμε λοιπόν είναι να υπάρχουν ή να υπάρχουν οι βασικές προϋποθέσεις για ένα δίκαιο εμπόριο, για δίκαιες συναλλαγές να ισχύουν και στο εσωτερικό της Ένωσης και στο εξωτερικό για τις εξαγωγές τα ίδια πράγματα και αυτό θα, σε αυτό θα επιμείνουμε και στο μέλλον. Watson. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η προηγούμενη συζήτηση ήταν για την πείνα και οι δυο συζητήσεις που κάνουμε εδώ όμως συνδέονται μεταξύ τους και η κυρία Επίτροπε δικαίως ζητούμε υψηλά επίπεδα στην ποιότητα του κρέατος αλλά για να παράγει κανείς ένα κιλό κρέας χρειάζεται κανείς 100 φορές παραπάνω νερό από ότι για να παράγει ένα κιλό σόγια. Θα πρέπει να πάψουμε να τρώμε κρέας. Θα πρέπει... Όπως είπε ο Chris Davis στην περασμένη συζήτηση θα πρέπει να επιμείνουμε οι πολίτες της Ένωσης να πάψουν να τρώνε κρέας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κώστιγκερ έχει το λόγο. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την ασφαλεία και την ποιότητα των ε, τροφίμων το θέμα είναι πολύ μεγάλο και όλα αυτά εξαρτώνται και από την προστασία των ζώων πέραν από αυτό που ελέγχθησαν και από την προστασία του περιβάλλοντος χρειάζεται να υπάρχει διαφάνεια από τον παραγωγό μέχρι το πιάτο αυτό όμως ισχύει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα των αγροτών μας και των κτηνοτρόφων μας θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να κάνουμε την ε, σχετική συζήτηση για να ορίσουμε τα πλαίσια με στα οποία μπορούμε να κινούμεθα και με τις τρίτες χώρες. Τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, ξέρετε πολύ καλά ότι η Ρουμανία δεν ε, μπορεί να πουλήσει χοιρινό κρέας ε, στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά μπορούμε να εισάγουμε από το 2010 χοιρινό κρέας από άλλα κράτη-μέλη και στη συνέχεια να τα εξάγουμε. Πρέπει να εφαρμόσουμε πολύ αυστηρούς κανόνες όσον αφορά το σφαγιασμό των ζώων και είμαι πεπισμένος ε, ότι οι κτηνοτρόφοι θα ήθελαν να αντικατασταθεί το σύστημα αυτό από ελέγχους ε, πιο, αυστηροί, πιο αυστηρούς ε, και από αφήσεις, αλλά θα έπρεπε να είναι οι κανόνες ήδη για όλους. έχει το λόγο τώρα. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame... Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε για την ε, παρουσίασή σας, η οποία μου φαίνεται ότι συνάδει με την ε, πολύ καλή σας δουλειά κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Ε, εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τον πληθυσμό μας. Οι συμπολίτες μας είναι έτοιμοι να δίνουν 100 ευρώ το κατέτος αν, αν μπορούμε να τους εξασφαλίσουμε την ποιότητα της διατροφής τους τη, λάβαμε γνώση της έκθεσης του ΦΑΟ και πρέπει να σας πω ότι εγώ πάρα πολύ δυσαρεστήθηκα βλέποντας πόσο ενοχλήθηκαν οι συνεργάτες σας, οι οποίοι προφανώς δεν μπορούσαν να απαντήσουν, δεν ήθελαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις μας. Θα έπρεπε να ντρεπόμαστε το να έχουμε, τόσο πολύ. Ε, ε, ε θα να, έχουμε, να ντρεπόμαστε που έχουμε αυστηρού κανόνε για να προστατεύουμε του καταναλωτέ μα και για όλου όσου θα θρέψουν του καταναλωτέ μα. Ε, ε, αυτές οι ίδιες ε, χώρες ε, που για παράδειγμα παράγουν αεροπλάνα μας επιβάλλουν κάποιες συνθήκες. Οι συνθήκες πρόσβασης της αγοράς είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί ακριβώς αφορούν τη διατροφή, αφορούν την υγεία των καταναλωτών μας και δεν πρέπει να, δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για αυτούς. Και τελευταίος ο μιλητής, ο κύριος Chcemy eksportować Ευχαριστώ. Κάποιοι θέλουν να εξάγουν και εμεί θέλουμε να εισάγουμε το εμπόριο. Είναι βασικό στοιχείο του σημερινού μας κόσμου. Αλλά βεβαίως πρέπει να τηρούνται κάποια πρότυπα και κάποια ασφάλεια και κάποια ποιότητα, με συγχωρείτε, η Ευρώπη για να διατηρήσει την ασφάλεια των προϊόντων που εξάγει και που εισάγει. Ε, έχει θεσμοθετήσει ελέγχους ε, κατά τους οποίους ελέγχεται ο σεβασμός κάποιων προτύπων. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται και στις εξαγωγές και στις εισαγωγές. Αλλά από ό,τι ακούσαμε κυρία Πρόεδρε, κάτι, ε, δεν είναι έτσι τα πράγματα πράγματα δεν, ενώ περιμένουμε να η να είναι οι και για τα εισαγόμενα προϊόντα αυτό δεν ισχύει κατάλαβα καλά η Ρωσία ή άλλες χώρες δεν επιβάλλουν και στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχους Ο λόγος σε εσά τώρα για να κλείσετε αυτή την πλούσια συζήτηση. Ευχαριστώ. Αξιότιμη μέλη, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το εξής. Αυτό που είπα δεν είναι ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κανόνες στις τρίτες χώρες και λυπούμε που μετά από μια δεκάλεπτη ή δεκαπεντάλεπτη παρουσίαση δεν σας έπεισα. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι ενώ εισάγουμε κρέας από τρίτες χώρες σήμερα από τη Βραζιλία εισάγουμε μην ξεχνάτε 5% των όσων των αναγκών μας σε βόλιο κρέας όσο λοιπόν εισάγουμε εξάγουμε κιόλα. προς τη Ρωσία και άλλους ένα δις το χρόνο είναι οι εξαγωγές μας στη Ρωσία ιδιαίτερα από την Ιρλανδία και προσπαθούμε να πείσουμε τη Ρωσία ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε τους κανόνες που εκεί ισχύουν. Γιατί εμείς θέλουμε να ισχύουν ισοδύναμοι αλλά όχι ταυτόσιμοι κανόνες. Έτσι λέει ο ΠΟΕ. Και αυτό κάνουμε. Ο λόγος για τον οποίο εφαρμόζουμε αυτούς τους κανόνες ασφαλείας στην Βραζιλία είναι ακριβώς επειδή από τις, αποτελέσ... από τις αποστολές μας, από τις αποστολές της ΦΑΟ, ανακαλύψαμε ότι τα πράγματα δεν έχουν καλώσει και γι' αυτό εφαρμόσαμε αυτού του αυστηρού κανόνε και σα έδωσα τα αριθμητικά στοιχεία. Η τελευταία αποστολή στη Βραζιλία. Ναι, κατέδειξε προβλήματα. Αλλά σα προκαλώ να κοιτάξετε όλε τι εκθέσει μα. και συγκρίνετε τις με τις εκθέσεις μας στα κράτη-μέλη. Και εκεί θα δείτε ελλείμματα και εκεί θα δείτε προβλήματα τα οποία ζητούμε από τις αρμόδιες αρχές να επιλύσουν. Όπως ζητούμε και από τις αρχές της Βραζιλίας. Προβλήματα στη Βραζιλία. Προβλήματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Βραζιλία. Τρεις εκμεταλλεύσεις είχαν τεράστια προβλήματα. Οι αρχές της χώρας πήραν τα μέτρα τους, απέσυραν τις εκμεταλλεύσεις αυτές από το κατάλογο των διεπιστευμένων και άσκησαν δίωξη κατά αυτών που τις πιστοποίησαν. Και άλλες εκμεταλλεύσεις είχαν πρόβλημα με κινητικότητα, κίνηση, διακίνηση των ζώων από φάρμα σε φάρμα, που είναι πρόβλημα για την ανείχνευσιμότητα, και αυτοί αδιώχθησαν. Και είπαν οι Βραζιλιανές αρχές ότι θα κοιτάξουν, θα επαληθεύσουν τα στοιχεία της βάσης δεδομένων για να μην υπάρχει περαιτέρω πρόβλημα. Τώρα, οι αποστολές της ΦΑΟ αυτοί τη δουλειά κάνουν και γνωρίζουν ότι θα βρουν προβλήματα. Η δική μας υποχρέωση είναι να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Είτε είναι στα κράτη-μέλη είτε είναι σε τρίτες χώρες. Διότι η υποχρέωσή μας είναι έναντι του καταναλωτή μας. Και σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσουμε τις αποστολές στη Βραζιλία και σε άλλες τρίτες χώρες, ούτως ώστε όταν ανακαλύπτουμε προβλήματα να διορθώνονται. Παίζουμε το παιχνίδι λοιπόν με δίκαιους όρους. Και για τους δικούς μας παραγωγούς και για τις τρίτες χώρες. Έγινε μια παρατήρηση για τη Ρουμανία. Ναι, η Ρουμανία, όπως και η Βουλγαρία, αλλά και πολλά άλλα κράτη-μέλη, παλιότερα είχαν πρόβλημα με την πανόλη των χείρων. Τη βοηθήσαμε πολύ τη Ρουμανία. Και σας προκαλώ να το επαληθεύσετε αυτό ενώπιον της κυβέρνησής σας τι αρρωγή παράσχαμε για να υπερπηδήσετε το πρόβλημα. Και είμαι σίγουρη ότι η Ρουμανία θα μπορέσει να ξεκινήσει πάλι τις εξαγωγές κρέατος στο πολύ εγγύης μέλλον. Χάρη στη δική μας βοήθεια. Χάρη στη βοήθεια που εμείς παράσχαμε για την εξάλληψη της πανόλης των χείρων. Εν κατακλείδη αξιότιμα μέλη. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η πρώτη μας ευθύνη είναι έναντι του Ευρωπαίου καταναλωτού. Και θέλουμε να παίξουμε το παιχνίδι με δίκαιους όρους και με ισότιμο τρόπο προς όλους τους παίκτες. Στα πλαίσια του ΦΑΟ έχουμε αυστηρούς κανόνες, θα συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε και αν υπάρχει πρόβλημα θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Αλλά θα πρέπει να είμαστε να επαγρυπνούμε και να είμαστε αυστηροί. Τώρα, αν η τάδε ή η δίνα εκμετάλλευση είναι στον κατάλογο ή όχι, αυτό εξαρτάται από τις αρχές της Βραζιλίας που θα πρέπει να δαπανίσουν τα κονδύλια που πρέπει να δαπανίσουν για να είναι σε θέση να πιστοποιήσουν πιστά αν μια εκμετάλλευση πρέπει να είναι στον κατάλογο ή όχι. Αυτά και σας ευχαριστώ. Η επόμενη συνεδρίαση αύριο 5η 26 Νοεμβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 13 μετά το μεσημέρι και από τις 15 έως τις 17 με την ημερήσια διάταξη η οποία έχει δημοσιευτεί στο έγγραφο συνόδου και που φέρει τον ίδιο τίτλο καθώς και στο ίντρανετ. Έληξε η συνεδρίαση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλή σας.